Καλό όχι μόνο, ζητούσαν να υλοποιηθούν τα όνειρα και οι ελπίδες μιας γενιάς Αλγερινών που σήμερα αποτελούν το 45% του πληθυσμού κάτω των 20 ετών και έχουν αποκλειστεί από οποιαδήποτε διαδικασία πρόοδου και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Γι' αυτό, αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση και από τα θεσμικά όργανα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη είναι να μπορέσουμε να σεβαστούμε, να ακούσουμε και να δράσουμε στο πλαίσιο τη κρίση αυτή. Να σεβαστούμε του χιλιάδε, τα εκατομμύρια ειρηνικού διαδηλωτέ. Να ακούσουμε τα νόμιμα αιτήματα αλλαγή για μεταρρύθμιση, για ελευθερίε και δικαιώματα. Και να δράσουμε για να δώσουμε απάντηση και διέξοδο σε ένα καθεστώ που χρειάζεται δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει ε, και για να απαντήσουμε στα αιτήματα του λαού τη Αλγερία. Σας ευχαριστώ κύριε Λόπες. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιλάν Μόν. Ευχαριστώ. Η Αλγερία είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και ζει σε μια κρίσιμη στιγμή. Ξέρουμε ότι έχει περάσει από μια δύσκολη περίοδο τη δεκαετία του 90 όταν ε, είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Ε, τώρα κλείνει άλλο στάδιο ε, υπό την Προεδρία του Μπουτεφλίκα που τίθεται τέλος και ήρθε η στιγμή για μια νέα ε, πολιτική περίοδο. Είναι σε μεταβλητική περίοδο Αλγερία και αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι ταχεία στο χρόνο και ε, θα πρέπει να είναι μια διαδικασία συμμετοχική μια αλλαγή ε, που πρέπει να έρθει καθώς ε, τη ζητούν ε, οι άνθρωποι με ειρηνικό τρόπο στο δρόμο και θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν θέλουν βία ούτε να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα οι Αλγερινοί ούτε θέλουν να ταξιδέψουν στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος γιατί θέλουν να κερδίσουν το μέλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους Αλγερινούς προσφέροντας τη συνεργασία μας αν την επιθυμούν ε, και με έναν ε, τρόπο δημοκρατικό και ειρηνικό ε, θα αποφασίσει ο ίδιος ο λαός το μέλλον του. Σας ευχαριστώ κύριε Μιγιανμόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Φρόιντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έγινε πολλής λόγος για την Αλγερία. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και χρόνια λέω ότι η Συρία δεν θα είναι η τελευταία χώρα που εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση αποτύχαμε η Αλγερία, ε, θα συναντήσουμε και την Αλγερία, θα τη βρούμε μπροστά μας σαν ε, αποτυχία. Η Αλγερία βράζει σαν ε, ένα καζάνι υψηλή πίεση, κάποια στιγμή θα εκραγεί. Και τι κάνουμε εμείς, κοιτάμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Στην Αλγερία υπάρχουν 40 εκατομμύρια κάτοικοι. Εάν ε, εδώ και κάποια χρόνια είχαμε μια ισχυρή και συνειδητή εξωτερική πολιτική και αν είχαμε χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά τη Συρία. Γι' αυτό η έκκλησή μου προς το Παρίσι, ε, ε, το Βερολίνο, τη Βιέννη και τη Στοκχόλμη να αλλάξει εξωτερική ε, πολιτική. Η, στην περίπτωση αυτή οι πολίτες στην Αλγερία αλλά και εδώ στην Ευρώπη θα μας ευχαριστούσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ξεκινήσω τη διαδικασία για το ΚΑΤΣΔΙ. Έχω λάβει τρία αιτήματα, θα τα δεκτώ όλα, ξεκινώντας από τον κύριο Ποσπισίλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα όλη τη συζήτηση με μεγάλη προσοχή. Εμείς έχουμε εκφράσει την πολιτική μας θέση και αυτό είναι θετικό. Πρέπει να ενισχύσουμε την διαδικασία εκδημοκράτησης της Αλγερίας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να φύγει ο πρόεδρος Μπουτεφλίκα. Από την άλλη, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει βία κατά τη μετάβαση αυτή. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την Αλγερία να διοργανώσει τις προεδρικές εκλογές με σκοπό να είναι μια ελεύθερη εκλογική αναμέτρηση, ε, συμπεριληπτική και να είμαστε προσεκτικοί όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. για να μην τεθεί κάποιο τέλος ε, στη διαδικασία εκδημοκράτηση. Κύριε Αγκόμες. Η Ευρώπη είναι η τα της ε, για τις σειράξει ε, στη Δυτική Σαχάρα και δεν μπορεί τώρα να έρθει εδώ και να προσποιείται ότι δεν βλέπει τι συμβαίνει στην Αλγερία. Είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να δει ότι ο λαός της Αλγερίας βγαίνει ειρηνικά στους δρόμους κατά μιας πέμπτης θητείας, κατά της μούμιας του Μπουτεφλίκα, κατά της στρατιωτικής εξουσίας υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Και δεν μπορούμε να είμαστε σιωπηλοί και να προποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε πρέπει να πούμε στο λαό ότι τον υποστηρίζουμε στην απέτησή του για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Ε, τα μήνυματα που θα στείλει η Ευρώπη μπορεί να είναι αποφασιστικά ε, ακριβώς ε, για να μην ε, συμβούν αυτά που έγιναν σε άλλες χώρες με την αραβική άνοιξη τα τελευταία χρόνια. Πρέπει οπωσδήποτε να υποστηρίξουμε το νέο λαό τη Αλγερία ε, στα αιτήματά του για τη δημιουργία θέσεων εργασία και η ευημερία του έχει να κάνει με τη δική μα ε, ευημερία και το ίδιο ισχύει και για την ασφάλειά του. Έχει να κάνει και με τη δική μα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριο ε, Φαριά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, παρά την ε, ε λαϊκή που ξεκίνησε και είχε ως ε, αποτέλεσμα να μην αναθεωρήσει, να ανανεώσει τη θητεία του ε, για πέμπτη φορά φλίκα ε, η αναστολή των εκλογών που ήταν προγραμματισμένη στις 28 Απριλίου ουσιαστικά σημαίνει ότι παρατείνεται η θητεία του και πάρα πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να διαδηλώνουν. Αν ενεργοποιηθεί το άρθρο 102 του συντάγματος ε, που προβλέπει την καθαίρεση του Προέδρου όπως προτείνουν κάποιοι στρατιωτικοί τώρα, ε, το κίνδυνος μπορεί να να επιταθεί και να υπάρχει αστάθεια σε όλη την περιοχή και αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες και την Ευρώπη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της παράνομης μετανάστευσης. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει όλες τις δυνάμεις που θα οργανώσουν ελεύθερες εκλογές πολύ σύντομα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα νέο επεισόδιο σαν αυτά που είδαμε στην Αραβική Άρξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Adesso la parola. Και τώρα, το λόγο έχει ο Επίτροπο Φαν, εξ ονόματος της ΥΠΑΤΗΣ εκπροσώπου εξωτερικών υποθέσεων και πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Um, στο πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Αλγερία που είναι ένας εταίρος, ε, μα ένας εταίρος μας κλειδί στην ε, περιοχή του Νότου. Ε, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η, να προσεγγίσουμε την ε, κατάσταση με όρους νομιμότητας του παρόντος καθεστώτος. Εδώ δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ε, τωρινή διαδικασία. Θα πρέπει να το κάνουμε όταν οριμάσουν οι προϋποθέσεις. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τα διάφορα βήματα που γίνονται και θα πρέπει να τονίσουμε ότι απόκειται στον αλγερινό λαό να αποφασίσουν για τον τρόπο που θα γίνει η μετάβαση αυτή. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή που δίνετε σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα και να σε ευχαριστώ και την επαγρύπνησή σας. Ε, ευχαριστώ με πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Τώρα στην μεσή διάταξη έχουμε τη δήλωση τη Πρόεδρου τη Επιτροπή Επίτευξη Προσώπου τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια για τα πέντε έτη παράνομη κατοχή τη Κρυμαία από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Ιωάννης Χάν. Πάντοτε εκπροσωπώντας την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, είπε την πρόσωπο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πριν πέντε χρόνια η Ρωσική Ομοσπονδία παράνομα προσάρτησε ένα μέρος της Κρυμαίας και την ε, Σεβαστούπολη. Για πέντε χρόνια μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την εδευκή κυριότητα της Ουκρανίας και την εθνική της κυριαρχία. Δεν αναγνωρίζουμε, ούτε θα αναγνωρίσουμε αυτή την παραβίαση του διεθνούς ε, δικαίου. Παραμένουμε στην πολιτική μας για τη μη αναγνώριση. Η επιδείνωση της ε, κατάστασης ε, στην περιοχή προκαλεί ανησυχίες με αυξανόμενη θετικοποίηση της Χερσονήσου και το περασμένο Νοέμβριο με το επεισόδιο που είδαμε ε, μας ε, υπενθύμησε τον αρνητικό αντίκτυπο της προσάρτησης στην ε, περιφερειακή σταθερότητα. Περιμένει η Ένωση από τη Ρωσία να απελευθερώσει τα μέλη του πληρώματος και τα σκάφη που τέθηκαν υποκράτηση εκείνη τη μέρα. Θα πρέπει να σεβαστεί τα δικαιώματα της ε, εκπροσώπησής τους από τις ε, προξενικές αρχές. Περιμένουμε από τη Ρωσία να τους χορηγήσει και την απαραίτητη ιατρική περίθλιψη. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση επίσης πηγάζει από την κατασκευή της ε, γέφυρας Κέρτς χωρίς την έγκριση της Ουκρανίας. Πριν λίγο καιρό η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει ένα καθεστώς εποπτείας που περιορίζει την ναυσιπλοεία από και προς τους λιμένες της Κρυμαίας και πολλά σκάφη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, υποφέρουν από καθυστερήσεις μπορεί να διαρκέσουν πολλές ημέρες. Περιμένουμε από τη Ρωσία ε, να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Κέρτς ε, προς και από τη θάλασσα του Αζόφ σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Καλωσορίζουμε την προσέγγιση της Ουκρανίας να ζητήσει δικαιοσύνη όπως ε, συμβαίνει δυνάμει της σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης προσάρτησης. Ε, ε, λυπούμαστε και για τον ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη Χερσόνησο και κυρίως ε, τα δικαιώματα των Τατάρων έχουν παραβιαστεί. Έχουν ε, κλείσει μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι δραστηριότητες του Μετλής έχουν απαγορευτεί και διώκονται μέλη της κοινότητας. Θα συνεχίσουμε να καλούμε για την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση του Όλεφ Σέντσοφ που έλαβε πέρσι το βραβείο Σαχάροφ και υπάρχει και φωτογραφία του εκτός, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυμίζει στους ανθρώπους ε, ε, την υπόθεση αυτή. Επίσης καλούμε για την απελευθέρωση πολλών άλλων όπως ε, την Αλεξάνδρα Κοσένκο, τον Αντάν Πενκεύκο, τον Νικόλα Σέμενα, τον Βολτιμίρ Μπάλοκ και τον Εμίρ Χουσέιν Κόκο που είναι υποκράτηση και έχουν καταδικαστεί στη Ρωσία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ε, καλούμε να διορθούν όλες οι περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ε, να υπάρχει πρόσβαση στη χερσόνηση της Κρυμαίας. Επίσης, δυστυχώς συνεχίζουμε να βλέπουμε παραδείγματα Ουκρανών πολιτών που παράνομα κρατούνται στη Ρωσία. Ο Παύλο Ρίπ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση πρόσφατα και επίσης αναμένουμε να απελευθερωθεί. Επίσης αδράτουμε κάθε ευκαιρία για να θέτουμε με μονομένες ε, περιπτώσεις δημόσια και δημερός με τους Ρώσου ομολόγους. Ε, η Ουκρανία δεν είναι μόνη της απέναντι στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Έχουμε σταθεί δίπλα στον εταίρο μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Καταδικάζουμε την ε, κατασκευή της γέφυρας Κέρτς ε, και καταγγέλουμε την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στον Εύξηνο Πόντο και στη θάλασσα του Αζόφ. Η θέση μας για την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και της Σεβαστούπολης έχει επαναληφθεί πολλάκις Κυρίω στι δηλώσει τη ΥΠΑ εκπροσώπου εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι 17 Μαρτίου. Ε, αναφέρθηκε δημοσίω σε αυτό το θέμα και στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίση, λάβαμε μέτρα για να δείξουμε στη Ρωσία ότι έχουν κόστο οι δράσει της στι 15 Μαρτίου. Ε, ε, καταρτήσαμε έναν περιοριστικό κατάλογο για Ρώσους πολίτες που είχαν εμπλακεί στην άσκηση εξουσία στα στενά του ΚΕΡΤ στο Νοέμβριο. Η απόφαση αυτή λήφθη ε, παράλληλα με παρόμοιες ε, ανακοινώσει που έγιναν από του διατλαντικού εταίρου και έτσι δείχνουμε την ενότητά μας. Επίσης εντοπίσαμε περαιτέρω τομεί για περαιτέρω στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την Ουκρανική περιοχή που πλήττεται από το καθεστώ παρακολούθησης στη θάλασσα του Αζόφ. Εξετάζουμε να αναπτύξουμε συνδέσει με σιδηρόδρομο και με δρόμους, να υποστηρίξουμε τι μικρέ και επιχειρήσει επιχειρήσεις που ε, στοχεύουν στο να διαφοροποιήσουν ε, την ε, βιομηχανική δομή της περιοχής αυτής. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή χάλιβα εκεί. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε αμφιβολία για τη θέση μας, για το που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, στο πλευρό της βασικής αρχής, ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία και σημαντικότερα είμαστε στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας. Εμείς έχουμε επενδύσει στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο και ξέρει η Ουκρανία ότι η υποστήριξή μας θα είναι μόνιμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Να ξεκινήσουμε με τις πενευές εξονομητές των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μπρόκ από το ΕΛΚ. Για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Χάν, για την παρέμβασή σας και την σαφήνεια που είχε. Στο Ελσίνκι διατυπώσαμε ως Ευρωπαίοι δύο βασικές αρχές την ε, κυριαρχία μιας χώρας και τη δυνατότητα να αποφασίζει ελεύθερα με, ποιον, ε, με ποια χώρα δημιουργεί συνασπισμούς. Ε, ε, το δεύτερο είναι η σταθερότητα των συνόρων που δεν μπορούν μονόπλευρα να αλλάξουν. Και τις δύο αυτές αρχές παραβίασε η Ρωσία. Ε, κατέλαβε ένα τμήμα μιας ξένης χώρας, ένα άλλο τμήμα έκανε πόλεμο και στην Αζωφική προσπαθεί επίσης να αλλάξει την κατάσταση παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Ε, αυτή είναι από το 1945 η πρώτη ε, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν θα ε, πρέπει να γίνει ε, συνηθισμένη πρακτική στην Ευρώπη του 21ου αιώνα να παραβιάζονται κατάφορα οι αρχές αυτές. Θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην επιβολή των κυρώσεων οι, οποίοι, οι οποίες είναι και προς του ρωσικού λαού γιατί θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου. Ο πληθυσμός του, της Ουκρανίας σε ένα διποψήφισμα το 1991 ε, αποφάσισε την ε, του 90 αποφάσισε την ενότητα της Ουκρανίας και επίσης ε, αποφάσισε μια ευρωπαϊκή λύση να προσχωρήσει στην Ευρώπη. Ω εκ τούτου δεν υπάρχει απολύτω καμία νομοποίηση για τη Ρωσία να εγείρει άλλε αξιώσει που επικαλούμενοι ότι ο πληθυσμός της Ουκρανίας έχει καταπιεστεί. Ο Στάλιν είναι αυτός ο οποίος ε, καταπίεσε τους Τατάρους της Κρυμαίας. Αυτό θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα κατά νου και θα πρέπει με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίσουμε την ε, κατήσχηση του διεθνούς δικαίου στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών, το λόγο έχει η κυρία Γκόμες. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Η παράνομη κατοχή της Κρυμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία παραβιάζει κατάφορα την ε, διεθνή συνθήκη ε, του 1994 και επίσης παραβιάζει τα δικαιώματα του λαού της Ουκρανίας αλλά και των Τατάρων. Ο Πούτιν θέλησε ε, μια Ρωσία που δεν σέβεται τα ανθρωπίνα δικαιώματα και, δημιουργεί, και χρησιμοποιεί την Κρυμαία ε, με αποτρεπτικό τρόπο για τις ε, γειτονικέ χώρες. Ε, το ίδιο ισχύει και για τη Γεωργία. Έχουμε παράνομα κατεχόμενα εδάφη από τη Ρωσία και φυσικά ε, δεν διστάζει να αυξήσει την ένταση στον Αυξηνοπόλο και στην Αζωφική θάλασσα, αλλά και στη Βαλτική και μάλιστα θέλει να καταστρέψει την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν δεν αρκούν πολιτικές δηλώσεις, ούτε καν οι κυρώσεις αρκούν. Θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της στρατηγικής άμυνας της Ευρώπης, των πολιτών και όλων των κρατών μελών, γιατί η ένοπλη σύραξη είναι πραγματική, θα μπορούσε να ξεσπάσει και θα μπορούσαμε να έχουμε και πυρηνική καταστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο. Μην με αναγκάσετε να σας αφαιρέσω το λόγο, γιατί δεν επιθυμώ να το κάνω τώρα εξ ονόματος ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος Γιούρο για ένα λεπτό. Πρόσε. Ε, το ε, από την προσάρτηση της Κρυμαίας έχουν παρέλθει πέντε χρόνια. Η ασφάλεια της Ρωσίας δεν πέστη καμία αρνητική επίπτωση. Η Ευρώπη δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ε, το θα πρέπει ε, Καταρχήν ε, με το Nord Stream θα απομονωθούν οι, οι χώρες της Βαλτικής και κατά δεύτερο λόγο θα απομονωθεί και η Ουκρανία. Ε, ε, εμείς η Ευρώπη ε, προσπάθησε με την επιβολή κυρώσεων να δείξει τη δυσαρέσκειά της, αλλά δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ισορροπία. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια, πράγματι μια κοινή εξωτερική πολιτική. Ε, θα, δεν ε, μπορέσαμε να επιδείξουμε καμία έμπρακτη ελεγγύη, αλλά περιοριστήκαμε στα λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Από το Άλντε, ο κύριος Σελίμωβιτς για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την παράνομη ε, κατοχή της Κρυμαίας και τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχουμε σταθεί το, στα ύψη των περιστάσεων. Δεν ξέρω γιατί. Επειδή χρειαζόμαστε το ρωσικό φυσικό αέριο, επειδή φοβόμαστε τη Ρωσία. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα αντιδρούσαμε αν αυτό συνέβαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αξιότιμοι συνάδελφοι από τις χώρες της Βαλτικής μπορούν ε, να είναι 100% σίγουροι ότι σε περίπτωση επίθεσης θα τους προστατεύσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς αυτή τη θέση θέλει να μας βάλει το Κρεμλίνο. Να αρχίσουμε να αμφισβητούμε τη δυνατότητα να προστατευτούμε, να μας ε, προκαλέσουν, να μας διχάσουν. Επομένως, να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε μία ολοένα και πιο επιθετική Ρωσία. Γεωργία, Ανατολική Ουκρανία, Κρυμαία, μας δείχνουν πέραν πάσης αμφιβολία ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει ε, καμία δεύτερη σκέψη στο να αλλάξει τα σύνορα στην Ευρώπη εάν μπορεί. Και αυτό μας ε, αφήνει μόνο μία επιλογή, μόνο μία λύση. Πρέπει να δράσουμε από κοινού και αποφασιστικά. Οποιαδήποτε άλλη απάντηση, ε, κάποια διαπραγμάτευση, διαβούλευση ε, από το Κρεμλίνο εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποστείλουμε ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα. Ως εδώ, ήδη έχετε πάει παραπέρα από ό,τι θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να ασκούμε πιέσεις, να αποχωρήσει από τις κατεχόμενες περιοχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εξ ονόματος των Πρεσίνων Ευρωπαϊκής Ελευθερή Συμμαχία, η Αντιπρόεδρο Χαουτάλα, για ένα λεπτό παρακαλώ, Χάιντι. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη εκπρόσωπο που ε, τόσο απερίφραστα κατήγγειλε την παράνομη κατοχή της Κρυμαίας και είναι πολύ σημαντικό που πέντε χρόνια αργότερα μιλούμε ανοιχτά για αυτή την ε, ε, υπόθεση γιατί καταπιέστηκαν και παραβιάστηκαν τα δικαιώματα πολλών ανθρώπων και πολλοί νιώθουν ε, ότι τους έχουμε εγκαταλείψει. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να καταγγέλουμε ε, την προσάρτηση της Κρυμαίας και την παραβίαση των ε, πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τότε που υπήρξε αυτή η δυσμενής εξέλιξη. Πρέπει να έχουμε πάντα ειδική μνήμα για τον Όλεξ Έντσοφ, στον οποίο επανεμήθηκε το βραβείο Σαχάροφ και να ζητήσουμε ε, την ανεφόρον απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Μετά την προσάρτηση έχουμε και την ε, υιοθέτηση ε, μία σειράς νόμων που περιστέλουν την ελευθερία έκφραση στην Κρυμαία. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε και τώρα εξ της ΓΚΟΕ. Ευρωπαϊκή Ενωτική και Αριστερά των Πράσινων Χωρών. Παρακαλώ, Κουσουπερμού, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε τα πέντε έτη της κατοχής της Κρυμαίας, όπως το αποκαλείται, και νομική, όπως ο Μπρέχαν Μπρέφεν, μέλος του Συμβουλίου Ηθικής της Γερμανίας, το αμφισβητεί. Για όσους θυμόμαστε, ξεκινά όλη η διαδικασία με το Μαϊντάν και με την επέμβαση κάποιων κομμάτων αυτού του Κοινοβουλίου. Στη διαδικασία όμως ξεκινούν όλα πολύ πιο πίσω. Κρίμα που δεν μιλάμε για τα 20 χρόνια της επίθεσης του ΝΑΤΟ στη Ιουκοσλαβία για πώς τότε παραβιάστηκε το διεθνές δίκαιο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κατηγορούν κάποια σήμερα τη Ρωσία. Έγιναν πολλά λάθη κατά τη διάρκεια και μετά από αυτό η πολιτική κυριώσεων κατά της Ρωσίας και η απάντηση που κόστησε χιλιάδες θέσεις εργασίας σε Ισπανία και Ιταλία. Επίσης, ε, ε, τότε να χρησιμοποιηθούν ε, τα μέσα ε, μαζικής ενημέρωσης ε, διαδίδοντας προπαγάνδα ή χρησιμοποίηση ναζί όπως είναι ο Ρωμάν Σουχέμοβιτς. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα εξ ε, του ΙΕΝΕΦ, ο συνάδελφος Σαφχάουσερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το οποίο αρνείστε στην Κρυμαία το εκχωρείται στους ε, Κωσοβάρους. Καταγγέλλεται τους ε, Ρώσους, αλλά αναγνωρίζετε το Κωσυφοπαίδιο Καταγγέλλεται τους ε, Ρώσους, αλλά εγκρίνεται τον παράνομο πόλεμο του ΝΑΤΟ στην Ιουγκοσλαβία. Καταγγέλλεται το δημοψήφισμα στην Κρυμαία, αλλά υποστηρίζεται την παράνομη δήλωση ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου το 2008 η οποία παραβίασε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, ε προκυρήσετε, τίθεστε υπέρ του διεθνούς δικαίου αλλά στηρίζετε το Κωσυφοπέδιο. Ε, αυτό το οποίο μισείται στην, ε, στους πολίτες εκεί είναι η βούλησή τους να ενταχθούν στην ιστορική τους πατρίδα την ε, Ρωσία. Στο παρελθόν δόθηκε η Κρυμαία από τους Μπολσεβίκους ε, ε, ε, δόθηκε στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Πόλτσακ. Τη δέχεστε. Εγώ περίμενα να ακούσω ακριβώς τι θα πείτε, γιατί ακούω κάποιον ε, να μιλάει ρωσικά. Πιστεύετε ότι είναι αντικειμενική η κατάσταση αυτή. Η Ρωσική Τράπεζα έδωσε ένα δάνειο 10 εκατομμυρίων στο πολιτικό σας κόμμα. Γνωρίζετε το memorandum του 1994 όσον αφορά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στην περίπτωση αυτή. Δεν θα απαντήσω. Έχουν γίνει έρευνες. Όλα αυτά έγιναν με απολύτως ε, νόμιμο, κανονικό τρόπο. Ε, τα επιτόκια είναι 6%. Ε, παραπάνω από αυτό που θα έδινε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αυτό το οποίο είναι σκανδαλώδες είναι ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία τράπεζα να τους χρηματοδοτήσει. Και αυτή είναι, αυτές είναι μπολσεβίκικες ε, μέθοδοι. Υπάρχει μια άλλη κάρτα, μπλε κάρτα από τον κύριο Πρέντα. Παρακαλώ. Oui, monsieur, monsieur. Κυρία Σαφχάουσερ, έχω κάτι που προκαλεί περιεργία. γιατί σας βλέπουμε εδώ και πέντε χρόνια να υποστηρίζετε με πάθος όλες τις θέσεις του Κρομλίνου. Αυτά τα πέντε έτη υπήρχε μία θέση του Πούτιν και του καθεστώτος τους που δεν υποστηρίξατε. Πού να διαφωνείτε, έτσι μια μικρή ερώτηση. Με ένα μικρό ζήτημα, μια λεπτομέρεια ή 100% είστε μαζί με τον Πούτιν και με το Κρεμλίνο, να μας πείτε την αλήθεια. Αγαπητέ συνάδελφε, η πολιτική που υποστηρίζω είναι η πολιτική της Γαλλίας. Λυπάμαι. Δείτε τη θέση της Γαλλίας ε, κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Δείτε πως ο στρατηγός Ντεγκόλ ήταν ο πρώτος που επισκέφτηκε τη Ρωσία του Στάλι Δείτε πώς όλοι οι αρχηγοί κρατώ, του κράτους μας είχαν προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Δείτε και τι κάνει και ο πρόεδρος Μακρόν. Παρόλο που μερικές φορές δυσκολεύεται να τοποθετηθεί, η πολιτική της Γαλλίας πάντοτε ήταν μια ισορροπημένη πολιτική. Μια πολιτική ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας. Και ελπίζω έτσι να παραμείνει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σκέλαμ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε. Η βίαιη προσάρτηση της Κρυμαίας πριν από πέντε χρόνια αποτέλεσε παρα... κατάφορη παραβίαση της διεθνούς τάξης. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με την ε, επέμβαση του Χίτλερ στην Αυστρία πριν από 81 χρόνια. Ε, πράγματι, η βία η επίθεση δέχτηκε δρυμύτατη κριτική και ε, επιβλήθηκαν και κυρώσεις. Όμως, οι ε, διαφωνίες και η διάσταση απόψεων έχει μειώσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδαμε ότι είχαμε το σκηνικό με τους ναυτικούς πριν από μερικούς μήνες και το, μάλιστα και το πρόσφατο ψήφισμα κατά της Ρωσίας δείχνει ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση απειλή προς όλες τις γειτονικές της χώρες ε, στην Ευρώπη. Πρέπει να αποκαταστήσει η Ρωσία την ε, εδαφική ακαιρεότητα της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο συνάδελφος εσείς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πέντε χρόνια μετά την παράνομη κατοχή, της, την παράνομη κατάληψη Κρυμαίας από τη Ρωσία δεν μπορούμε παρά σε αυτό το κοινοβούλιο να καταδικάσουμε αυτή την παράνομη στάση της Ρωσίας. Όμως δεν μπορούμε παρά να την προσοχή και στις ε, φιλοπόλεμες συμπεριφορές ε, της χώρας αυτής ε, στα στενά του Κέρτσι και στη θάλασσα του Ασόφ καθώς και την αυξανόμενη ένταση στον Ευξηνοπόντα. Αυτό ζημιώνει όλη την περιοχή. Για όλα αυτά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως μια ερώτηση που πρέπει να θέσουμε εδώ είναι ξεκάθαρο. Η σημερινή Ρωσία δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Εγώ ήμουν και είμαι ε, αντισοβιετιστής. Όμως το να συγκρίνουμε τη Ρωσία με την Σοβιετική Ένωση ε, δεν είναι σωστό. Η δική μας θέση πρέπει να είναι επικριτική απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς που αμφισβητεί ε, και καταπατά θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα, τα οποία πρέπει να υπερασπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υποχρέωση να τα υπερασπίσει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ασής. Και τώρα ο κύριος Ντέμις Μάκερ. Yeah. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την ε, ξεκάθαρη θέση σας. Ε, η Κρυμαία είναι μια κλεμμένη χερσόνησο. Το 2014, για πρώτη φορά με τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, ε, επενέβη μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και προσάρτησε αυτά τα εδάφη. Τα πράσινα αυτά ανθρωπάκια ήταν Ρώσοι ε, έτσι. Ήταν μια πολύ καλά σχεδιασμένη στρατιωτική επιχείρηση. και έχει κλείσει μάλιστα η Ρωσία 47 ε, συμβάσεις. και το σύμφωνο της Βουδαπέστης ε, το 1994. Η κλεμμένη χερσόνησος αυτή, που παλιά ήταν τουριστικό θέρετρο, είναι μια μεγάλη στρατιωτική βάση με τις νέες ρωσικές προκλήσεις αυτό καθίσταται σαφές. Ο σεβασμός προς το διεθνές ε, δίκαιο είναι ε, θεμέλιος λήθος ε, της ειρήνης και της σταθερότητάς μας. Γιατί αν το αφήσουμε αυτό κατά μέρο, αμφισβητείται μετά και η δική μας ε, σταθερότητα και ειρήνη. Και αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρία Τζίλ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παράνομη κατοχή της ε, Κρυμαίας από τη Ρωσία διακινδυνεύει την ε, παγκόσμια ειρήνη. Κάτι το οποίο μπορεί πολύ γρήγορα να κλιμακωθεί σε μια ε, διεθνή απειλή για την ειρήνη. Και ο λαό τη Κρυμαία όλο ένα και περισσότερο απομονώνεται. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα οικονομικά συμφέροντα συνεχώ υπονομεύονται. Το Κοινοβούλιο έχει επανελειμμένως ζητήσει την ε, αποκατάσταση της εδαφικής κυριαρχίας και ενότητας και κυριότητας της Κρυμαίας. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η Ρωσία ε, χτίζει γέφυρες ε, και επιτίθεται σε σκάφη δεν φτάνει να δίνουμε βραβεία Σαχάροφ σε ανθρώπους όπως ο Όλεξ που αντιτίθενται σε αυτή την καταπίεση. Είναι σημαντικό αντιθέτω να αποστείλουμε ένα χειρό μήνυμα προς τη Ρωσία ότι το να αγνοεί κανείς το διεθνές δίκαιο έχει προεκτάσεις και συνέπειες. Και πρέπει να συνδράμουμε περισσότερο την Κρυμαία για την ασφάλειά τη. Πώ αυξάνουμε λοιπόν αυτή την πίεση προ τη Ρωσία, κύριε Επίτροπε, θεωρείτε ότι μπορείτε να πείσετε τα κράτη-μέλη να ε, ευθυγραμμιστούν και να στηρίξουν αυτό που είπατε προηγουμένω, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα η πρόεδρο Φωτίγα, για ένα μισή λεπτό παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Για πέντε χρόνια η και η Ομοσπονδία κατέχει παράνομα την ε, Κρυμαία και οι γεννήστες της Ιερσονήσου, η Τάταροι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο. Είναι το τρίτο κύμα παραβιάσεων κατά της κοινότητε αυτής. Το πρώτο ήταν το 1783 με την ε, μαζική ε, με το μαζικό διωγμό από το τσαρικό καθεστώς κατόπιν το 1945 ε, από το Στάλιν και πάλι είχαμε μαζική απέλαση του λαού της Κρυμαίας. Τώρα είναι μειονότητα στην Χερσόνησο και υφίσταται τεράστιες παραβιάσεις, παιδιά εξαφανίζονται, υπάρχουν πολιτικοί πρόσφυγες, υπάρχουν συλλήψεις, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φέτος, οι Τατάροι της Κρυμαίας ε, μαζί με όλη την Ουκρανία και ελπίζουμε όλη τη διεθνή κοινότητα ε, γιορτάζουν ε, την ε, επέτειο της τελευταίας τους απέλασης, του τελευταίου διωχμού. Χαίρομαι για τη δήλωσή σας, κύριε Επίτροπε, για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, προκειμένου να επιστραφεί και το έδαφος αυτό στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο η κυρία Γουόρτ για ένα λεπτό, παρακαλώ. Five Μετά χρόνια μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ενώνω τη φωνή μου με αυτό που καταδικάζουν την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η συνεχιζόμενη κατοχή της Χερσονήσου υποσκάφτει τη σοβαρά το κράτος δικαίου και τις διεθνείς σχέσεις. Ήδη έχω καταδικάσει εδώ τις ε, τρομερές ε, συνέπειες που έχει αυτή η κατάσταση στην πολιτιστική κληρονομιά στην Κρυμαία που συνεχίζει να καταστρέφεται επί τόπου με την απώλεια σημαντικών ιστορικών μνημείων. Εν τω μεταξύ, υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλλιτέχνε και άτομα τη πλειοψηφία συνεχίζουν να διώκονται στη Ρωσία και στα κατεχόμενα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιμείνει στο να ε, αρνείται να γνωρίσει την παράνομη κατοχή της ε, Κρυμαίας. Ε, ε, Ρώσοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις εκλογές και δημοψηφίσματα με την χρηματοδότηση κομμάτων της ακροδεξιάς. Εμείς θα συνεχίζουμε να περασπίζουμε το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις σχέσεις μας με τη Ρωσία αλλά και με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Πέντε αιτήματα για το λόγο. Και ε, έχουμε από το ΕΛΚ τα αιτήματα. Θα τα δεκτώ όλα, ξεκινώντας από τον κύριο Ποσπισίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα και ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε, η πλειοψηφία μας μάλλον ε, θεωρεί ότι η προσάρτηση της Κρυμαίας είναι μια παράνομη ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ότι η Ρωσία παρανόμως ε, συνεχίζει τις δραστηριότητες της και στη θάλασσα του Άσοφα για παράδειγμα. Μετά είναι και το ζήτημα των μυρωτήτων στην Κρυμαία. Πολύ σημαντικό και αυτό οι Τατάροι της Κρυμαίας, για παράδειγμα, πλήττονται ιδιαιτέρως, ε, καθώς και οι ακτιβιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και οι δημοσιογράφοι. Επομένω, δεν είναι μόνο το θέμα τη ε, παραβίαση του διεθνού δικαίου, αλλά και η αντιμετώπιση ε, του λαού τη Κρυμαία. που επιθυμούν να ζήσουν ανεξάρτητα από τη Ρωσία. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαρία, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρώτα. Πέντε χρόνια μετά τη βαράνου προσάρτηση της Κρυμαίας, ε, συνεχίζονται οι παραβίαση των ανθρωπικών δικαιωμάτων, κυρίως των τετάρων ε, και οι παράνομες ε, συλλήψεις στο Κρεμλίνο. Συνεχίζει να προωθεί τα σχέδιά του και μάλιστα ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία. Τώρα η ερώτηση είναι πώς σε άλλους επαιτίους θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ μέχρι η δαφική ακυρεότητα της Ουκρανίας να αποκατασταθεί και να γίνουν σεβαστές συμφωνίες του ΜΙΣ και η Ένωση θα πρέπει όχι μόνο να ανανεώσει τις οικονομικές κοινώσεις μέχρι, από τον, που ισχύουν μέχρι τον Ιούλιο, αλλά ε, θα πρέπει να καταπολεμήσει και το ξέπλυμα χρήματος από το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης. Ε, αυτό ε, θα πρέπει να γίνει μέσω της συμπερίληψης Ρουσίας στη μαύρη λίστα και στην ε, θέση διαδικασία επί παραβάση για τα κράτη που δεν έχουν ακόμα μεταφέρει στο ιστορικό τους δικαίωτη την τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δεν μπορεί να επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να δίνουν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες οξυγόνο στη Ρωσία με τον τρόπο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. κυρία Σόντροβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο Χάν ε, για την ε, σαφή του τοποθέτηση κατά της ε, ρωσικής στάσης στην Κρυμαία. Πέντε χρόνια λοιπόν έχουν περάσει από την προσάρτηση, αλλά συνεχίζει να μας τρώει αυτή η αδικία. Πέντε χρόνια λοιπόν έχουν ε, περάσει από την Ολομέλεια του ΟΗΕ που έλεγε ότι ήταν, είναι άκυρη η προσάρτηση της Κρυμαίας. Και ό,τι αφορά την ε, στάση της Ρωσίας απέναντι στον ε, κρεμεκό λαό, υπάρχουν παράνομοι διωγμοί, φυλακίσεις. Η μοίρα της Κρυμαίας εξαρτάται και από την στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Στέτινα, παρακαλώ. Ε, Κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, το Ιούνιο του 2000 επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Ρωσία. Το 2014 επίσης επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά Ρώσων πολιτών παρόλο που δεν είχαν άμεσο, άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία της ε, Ρωσίας παρόλα αυτά ε, θα μπορούσαν να είχαν έναν αντίκτυπο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε το Κοινοβούλιο για τα δικά του ε, συμφέροντα στην ε, Ουκρανία και η Άνω Βουλή ενέκρινε ομόφωνα αυτές τις αποφάσεις. Συστήνω λοιπόν να υπάρξει όξυνση αυτών των μέτρων ε, μέχρι και απαγόρευση εισχώρησης των μελών του Άνω της Άνω Βουλής της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πόλτσακ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. τα πέντε χρόνια της ε, κατοχής της Κρυμαίας σημαίνουν ε, πέντε χρόνια παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για το περβίαστο των συνόρων, αλλά καταπατάται και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίω των Τατάρων. Αυτοί είναι πολίτες χωρίς δικαιώματα. Η Ουκρανία χρειάζεται τη βοήθειά μας. Εγώ υποστηρίζω ε, πλήρως ε, τη συνεργασία Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να ζητήσω συγγνώμη ε, από το λαό της Ουκρανίας ε, για τις δράσεις ε, του Μίλος Ζάμαν, ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία για να ζημιώσει τις σχέσεις Τσεχίας-Ουκρανίας. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από τους Ουκρανούς πολίτες. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τις κυρώσεις και θα πρέπει να επιμείνουμε να επιστραφεί η Κρυμαία στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, πάντοτε, εξ ονόματος του Επιτροπή Επιτροπής τη Εκπροσώπου της Ένωσης, ε, το λόγο έχει Επιτροπος Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακολουθώντας την συντριπτική πλειοψηφία των ε, παρεμβάσεων, μπορούμε όλοι να συμπεράνουμε θα πρέπει να συνεχίσουμε τη μη αναγνώριση της ε, παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας και να δώσουμε στο θέμα αυτό μια προτεραιότητα παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς της εξελίξης στην ε, Ζωφική και εξετάζοντας πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, σε διμερές ή πολυμερές ε, επίπεδο για να καταγγείλουμε την παράνομη προσάρτηση της ε, Κρυμαίας. Και αυτή είναι η ομόφωνη τοποθέτηση όλων των χωρών μελών. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τον κύριο Πρέντα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα πολύγλωσσος. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Τώρα θα περάσουμε στην έκθεση Φέι Κατάσταση μετά την Αραβική Ένωση, μελλοντικέ ενέργειε για την περιοχή τη Μέση Ανατολή και τη Βορειά Αφρική. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ, Μπράντου. Ευχαριστώ. Πριν 8 χρόνια, χιλιάδε γυναίκε και άνδρες, ιδίω νέοι, βγήκαν ε, στις ε, πλατείες ε, σε όλη την νότια όχθη της Μεσογείου για να ζητήσουν περισσότερη δημοκρατία, το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών, δουλειά και κοινωνική ένταξη. Οκτώ χρόνια από εκείνες τις διαμαρτυρίες που σήμαιναν ένα σημείο ρήξης με τα συστήματα του παρελθόντος και κυρίως με την ε, δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε ε, ουσιαστικά με την Αραβική Ένοιξη μια σειρά ε, πολλών εξελίξεων που οδήγησε διάφορες χώρες σε νέα καθεστώτα ή και σε εμφύλιο πόλεμο. Ταυτόχρονα η Ευρώπη καταρχήν προσπάθησε να παρακολουθήσει τις ε, δημοκρατικές διεκδικήσεις που αναδύθηκαν. Όμως ε, στη συνέχεια επειδή αυξανόταν ε, η απειλή η τρομοκρατική από το ΆΕΣΙΣ και η κρίση του προσφυγικού, η Ευρώπη θέλησε να επικεντρωθεί στην σταθεροποίηση των χωρών, στη συγκράτηση της μετανάστευσης και έτσι λοιπόν επαναλάβαμε τα λάθη του παρελθόντος και δεν καταλάβαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ακολουθούσαμε το φαύλο κύκλο που προσπαθούν, από τον οποίο προσπαθούν να βγουν οι λαοί τη περιοχή. Και το διαβλέπουμε και στην Αλγερία σήμερα. και Κινδυνεύει να γίνει μια νέα Συρία, αν για μια ακόμη φορά υποτιμήσουμε την κατάσταση η Ένωση θα είχε πολλά μέσα στη διάθεσή της για μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική. Όμως μια ανανεωμένη δράση θα πρέπει να ξεκινήσει από μεγαλύτερη ενότητα και συντονισμένη προσέγγιση. Αν το κάθε κρατό μέλος συνεχίζει να επιδιώκει τα δικά του συμφέροντα, ε, βράχει πρόθεσμα, ε, τότε θα συνεχίσουμε να ε, μην μπορούμε να επηρεάσουμε την ε, κατάσταση στην περιοχή ε, και τελικά μόνο θα πληρώνουμε όπως έγινε στη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε την πολιτική μας προς ε, αυτή την πολύ σημαντική περιοχή στη γειτονία μας. Όπως είπαμε και στην συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική θα πρέπει να επενδύσουμε όχι απλώς σταθεροποίηση αλλά στην εφεκτικότητα των κοινωνιών το να υποστηρίζουμε αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά, όμως τελικά μπορεί αυτό να οδηγήσει σε έκρηξη. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιώματων, στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό που αναδύθηκε από την Αραβική Άνοιξη ήταν μεγάλη κρίση εμπιστοσύνη ε, από του πολίτε απέναντι στους θεσμού που ζητούν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Θα πρέπει η Ένωση να το υποστηρίξει αυτό. Προτείνουμε λοιπόν στην έκθεση μία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την άποψη των λαών, ένα συνεχή και διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών ε, και σε τοπικό επίπεδο. Μία προσέγγιση που να θεωρεί πρωταγωνιστές τους νέους ε, που είναι δυναμικό στοιχείο αλλά και ευπαθές αυτών των κοινωνιών. Γι' αυτό προτείνουμε να συστήσουμε σε αντιπροσωπείες της Ένωσης ε, γνωμοδοτικά συμβούλια των νέων ε, και προτείνουμε να υπάρξει και ένα ευρωμεσογειακό εράσμους και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να θέσουν τέλος στην πώληση όπλων ε, που χρησιμοποιούνται από καθεστώτα που δεν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναλαμβάνουμε επίση ότι μια μεγαλύτερη συνεργασία ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και δικαστική και αστυνομική συνεργασία. Έχουμε την περίπτωση Τζούλιο Ρετζένη, για το οποίο περιμένουμε ακόμα την αλήθεια. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν το παράδειγμα και πιστεύουμε ότι ε, με αυτή την έκθεση προωθούμε το διάλογο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία ε, με τους εταίρους μας ε, στην Μεσόγειο, στον νότιο τμήμα της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ τώρα. Εξ ονόματος της είπα εκπροσώπους και πάλι ο Επίτροπος Χάν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε μέλη. Πρώτα απ' όλα θα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Μπελιφέη, για την έκθεσή του για την κατάσταση σε ορισμένες χώρες της περιοχής ΕΜΕΝΑ μετά την Αραβική Άνοιξη. Συμφωνούμε αρκετά με τα βασικά στοιχεία της έκθεσης σχεδόν μια δεκαετία μετά από την Αραβική Άνοιξη. Πολλά από τα αιτήματα που οδήγησαν τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό ακόμα δεν έχουν απαντηθεί σε πολλές από αυτές τις χώρες. Ε, καλύτερες δημοκρατίες, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερία έκφρασης τελικά είναι το αίτημα για πιο συμπεριληπτικά συστήματα διακυβέρνηση. Αυτά βρέθηκαν στον πυρήνα τη Αραβική Άνοιξη. Πολλέ χώρε, κάποιε χώρε μάλλον, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπω η Τινησία, που αποτελεί ακόμα σημείο αναφορά για την περιφέρεια. Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική ξεκαθαρίζει ότι η σταθερότητα σε αυτή την περιοχή δεν μπορεί να διασφαλιστεί εάν ε, παρακάμψουμε ή αμελήσουμε αυτά τα αιτήματα. Για να έχουμε ανθεκτικό κράτο πρέπει να έχουμε μια ανθεκτική κοινωνία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε δημοκρατία, διαφανεί θεσμού, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Τι εξή παρατηρήσει έχω να κάνω. Πρώτον, κανεί δεν υποστηρίζει την κοινωνία των πολιτών σε αυτέ τι περιοχέ όσο εμεί οι Ευρωπαίοι. Όχι μόνο έχουμε θεσπίσει ε, Φόρουμ Κοινωνίας των Πολιτών για τον ε, γειτονικό μας Νότο, στο οποίο έχουν τεθεί επικεφαλής οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Αλλά βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών. Ε, εργαζόμαστε για την προώθηση συνεχών διαβουλεύσεων μαζί τους με τη βοήθεια συγκεκριμένων σημείων επαφής με κάθε αντιπροσωπεία. Αναφέρεται επίση στην έκθεση το θεμελιώδε έργο τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το έργο μας ε, σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των ε, υπερμάχων ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται και για τη συνεργασία μας με τους νέους. Καμία ανθεκτική δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την πλήρη για ενεργό συμμετοχή των νέων. Πρέπει να βρουν τη θέση τους λοιπόν και στην κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να ακούσουμε τις φωνές τους. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε μια ασφαλή πλατφόρμα για την ε, περιοχή αυτή για να, μας, ε, για να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Young Med Voices Plus ονομάζεται με σκοπό οι νέοι να έχουν έναν ανοιχτό διάλογο με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Πριν από ένα μήνα είχαμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στον διάλογο 5 συν 5 της ε, Δυτικής Μεσογείου και να διαμορφώσουμε από κοινού τα αποτελέσματα της συνάντησης. Ερχόμαστε λοιπόν σε επαφή με την κοινότητα των πολιτών σε όλα τα θέματα, ακόμα και στα πιο δύσκολα. Το δεύτερο λοιπόν που ήθελα να πω έχει να κάνει με τη Συρία. Έγινε λοιπόν προσφάτως η διάσκεψη για το μέλλον της Συρίας και αποφασίσαμε η κοινωνία των πολιτών της Συρίας να βρεθεί ε, στο επίκεντρο της ε, διάσκεψης. Πάνω από 400 ΜΚΟ συμμετείχαν λοιπόν ε, που δραστηριοποιούνται επιτόπου καθημερινά με ειδική εστίαση στις γυναίκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, γιατί η Συρία ανήκει στους Σύρους και ο μοναδικός τρόπος να δώσουμε τέλος αυτή την ε, σύραξη είναι να βοηθήσουμε τον λαό, να δημιουργήσουμε ε, μια νέα συμφιλειωμένη, ενωμένη Συρία. Ξέρουμε ότι η κατάσταση στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή δεν είναι ιδανική και οι φιλοδοξίες ε, της και τα όνειρα της Αραβικής Άνοιξης πολύ συχνά διαψεύστηκαν. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε ε, άοκνα την προσπάθειά μας με όλους τους ε, φορείς, με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και με τις κυβερνήσεις και να προωθήσουμε την αλλαγή που θέλουμε να δούμε σε αυτή την περιοχή. Το τελευταίο που θέλω να πω, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο των δικών μας προσπαθειών. Εμείς πάντα θίγουμε το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κάποιες φορές ε, δημοσίως, ε, κάποιες φορές κατηδίαν στις συναντήσεις μας με τους ομολόγους μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους φίλους μας στην άλλη όχθη της Μεσογείου να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες τους προς καλύτερες δημοκρατίες, περισσότερη ελευθερία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τα όσα έχετε κάνει, ακόμα και για την κριτική σας, την οποία λαμβάνουμε υπόψη και θα φροντίσουμε ε, να τη διασκεδάσουμε. Ε, κανείς ε, δεν μάχεται όσο μαχόμεθα εμείς για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την Μαρία Ρενά που θα έπρεπε να μιλήσει εξ νόμου της Επιτροπής Γυναικών. Αν έρθει θα της δώσω το λόγο. Θα δώσουμε τώρα το λόγο σε προσώπους των πολιτικών ομάδων για το ΕΛ και για ένα μισή λεπτό κύριος Μπροκ. σε.